Υπότιτλοι AUTHORWAVE <clears throat> Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάει η συνεδρίασή μα. Μία μεικτή συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης υπό την προεδρία της κυρίας Ζολή, της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Αντικαθιστώ τον πρόεδρο Αλμπερτίνη και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό την προεδρία της κυρίας Σωτά. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις για τα πρακτικά, θα μπούμε στην ουσία της σημερινής συνεδρίασης και θα ακούσουμε την παρουσίαση των υποψηφιωτήτων, ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσει σε ποιον θα χορηγήσει το βραβείο Ζαχάροφ. Υπενθυμίζω ότι κάθε χρόνο από εδώ και πλέον από 20 χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει αυτό το βραβείο, ούτω ώστε να ανταμείψει είτε προσωπικότητες είτε οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, καταπολεμώντας την ε, αδικία, την καταπίεση και που χάρη στην έγκλη τους και στην φήμη του γίνονται σύμβολο της δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. δίδοντας το βραβείο Ζαχάροφ, υπογραμμίζουμε κάποιες ε, σημαντικές δράσεις, την ελευθερία της ε, σκέψης και της ε, έκφρασης, την καταπολέμηση της, του μίσους και με αυτόν τον τρόπο εκφράζουμε την, θέληση, την άποψή μας ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες είναι όχι μόνο το δικαίωμα στη ζωή και η φυσική ακεραιότητα, αλλά η ελευθερία σκέψης και η ελευθεροτυπία που αποτελούν ένα από τα χαρακόμματα του αγώνα κατά της βίας, της ε, καταπίεσης και βασικό στοιχείο της ανοιχτής κοινωνίας και δημοκρατίας. Δίνω το λόγο στην ε, κυρία Ζολή, πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης, ούτως ώστε να πει και εκείνη δύο λόγια κατά την έναρξη των εργασιών μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω όλους σε αυτή την συνεδρίαση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, όπου παρουσιάζουμε τις υποψηφιότητες για το βραβείο Ζαχάροφ. Ξέρουμε στην καθημερινότητά μας ε, στη ζωή μας πόσο σημαντικά είναι τα σύμβολα. Και νομίζω ότι ο συμβολισμός αυτού του βραβείου είναι πάρα πολύ σημαντικός λόγω της ποιότητας των ε, υποψηφιωτήτων και των βραβείων που δόθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια. Φέτος, οι 7 τους 10 υποψηφίους, άτομα είτε οργανώσεις, προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για μια ουσιαστική ανάπτυξη των κοινωνιών μας. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ τις υποψηφιότητές μας, ούτως ώστε να διατηρήσουμε το συμβολικό χαρακτήρα του βραβείου. Με μεγάλη χαρά θα δώσω το λόγο στην κυρία Οταλά, που είναι η Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ την κυρία Ζουλή. Θα ήθελα εν ονόματι της δικής μου υποεπιτροπής να σας καλωσορίσω σε αυτή τη συνεδρίαση για την επιλογή του νικητή, καταρχάς των υποψηφιωτήτων των, του βραβείου Σαχάροφ. Θα παρουσιάσουμε όλες τις οργανώσεις και όλα τα πρόσωπα. Πριν από 20 χρόνια πέθανε ο Ανδρέη Σαχάροφ. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική χρονιά φέτος Συζητήσαμε πάρα πολύ για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Τον Δεκέμβριο, όταν δώσουμε το βραβείο, θα κάνουμε μία επίσημη εκδήλωση. Προς το παρόν, δεν έχουμε αποφασίσει. Αυτές οι προτάσεις έγιναν από τουλάχιστον 40 βουλευτές, είτε από πολιτικές ομάδες. Θέλω να το υπενθυμίσω αυτό. Και σε αυτή τη φάση οι ευρωβουλευτέ μπορούν να υποστηρίξουν μόνο μία υποψηφιότητα. Αυτό θέλω να το τονίσω, να το ξέρουν όλοι. Σε επίπεδο ομάδων, προέδρων ομάδων, επίσης θα πρέπει να υποδειχθεί μία οργάνωση ή ένα άτομο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δηλαδή, ανεξάρτητα αν η οργάνωση έχει ή δεν έχει νομική προσωπικότητα. Η Γραμματεία έλαβε 10 υποψηφιότητες με το κλείσιμο της προθεσμίας το Σεπτέμβριο. Οι 10 προτάσεις την χάνουν επεξεργασίας εξετάζουμε αν γίνεται σεβα... υπάρχει σεβασμός των κριτηρίων ε, με βάση τα όσα αναφέρονται στο κανονισμό του βραβείου. Σας υπενθυμίζω ότι έχετε μία περίληψη γραπτή για κάθε υποψήφιο. Άτομο ή οργάνωση. Και θα ήθελα να σας αναφέρω τις 10 αυτές προσωπικότητες. Θα ήθελα επίσης να δώσω το λόγο σε κάθε υποψήφιο να εκφραστεί για πέντε λεπτά το πολύ. Έχουμε τον ε, δόκτορα Ιζελντίν Αμπουελάης, το Ίδρυμα Βιντσέντε Φερέρ, τον Νταβίδ Ιζάκ, την κυρία Μαριάμ Λαμιζάνα, εν συνεχεία μια ομάδα ατόμων, Λουτμίλα Αλεξέγεβα, Άλεγ Ορλόβ, και Σεργέη Κοβάλεφ της οργάνωσης Memorial και όλους τους υπόλοιπους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Εν συνεχεία, έχουμε την ίδια την οργάνωση Memorial. Σε συνδυασμό με αυτές τις δύο προτάσεις, θα ήθελα να σας πω ότι τα άτομα τα οποία παρουσίασαν αυτούς τους υποψήφιους θα πρέπει να βρουν μία λύση μέχρι την επόμενη εβδομάδα όπου θα αποφασίσουμε ε, για ένα short list τριών υποψηφιότητων. Εν συνεχεία έχουμε τον ε, δόκτωρα Ντένις Μουκουβέγγε, εν συνεχεία τον ε, εδεσιμότατο Θαδέους Νγκιέν Βαν Λί και άλλες δύο υποψηφιότητες, Σάντι Σάντρ, εξ ονόματος της Νέντα και τελευταίο τον Ρομπέρτο Σαβιάνο. Έχουμε αυτούς τους 10 υποψήφιους. Ε, δίπλα στο όνομά τους έχετε την περίληψη. Μπορώ να δώσω βεβαίως το λόγο σε οποιονδήποτε υποψήφιο είναι παρόν ή σε κάποιον που πρότεινε αυτά τα άτομα για να εξηγήσει την πρόταση. Με αλφαβητική σειρά λοιπόν. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δύο βουλευτές θα θέλουν, θέλουν να μιλήσουν για κάθε υποψήφιο. Ανά υποψήφιο υπάρχουν πέντε λεφτά συνολικά. Επομένως, σας παρακαλώ κοιτάξτε το ρολόι, κοιτάξτε το χρονόμετρο. Για κάθε υποψήφιο πέντε λεπτά συνολικά, επαναλαμβάνω. Θα ήθελα να δώσω το λόγο σε όσους πρότειναν τον δόκτορα Ιζελντίνα Μπουελάης. Κυρία Ντεκάιζερ, καταρχήν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η υποψηφιότητα του δόκτορα Ιζελντίν Αμπουελάης παρουσιάζεται από τον Hans Gert Πέτερινγκ, από το ΕΛΚΑ, από μένα και την Καρολίν Λιουκά εγώ θα μιλήσω για τον Hans Gert και για μεν, τον εαυτό μου και οι πράσινοι θα εξηγήσουν τη δική τους, τους δικούς τους λόγους. Θα ήθελα να σας πω ότι με κάθε ταπεινότητα θα ήθελα να μιλήσω ε, για την περίπτωση του δόκτωρα Μπουελάης, γιατί η περίπτωσή του είναι προφανής. Πρόκειται για ένα Παλαιστίνιο γυναικολόγο που δουλεύει στη λωρίδα της Γάζας. Ε, Κατά τη διάρκεια των ε, στρατιωτικών επιχειρήσεων, ο δόκτρος έχασε τις τρεις κόρες του μπροστά στις ε, κάμερες και η θλίψη του και οι φωτογραφίες από εκείνες τις στιγμές έκαναν το γύρο του κόσμου. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ο γυναικολόγος αυτός στη Γάζα δουλεύει επίσης και σε ένα Ισραηλινό νοσοκομείο. Και μετά τον τραγικό χαμό των παιδιών του συνέχισε να δουλεύει σε αυτό το νοσοκομείο στο Ισραήλ και, σε... και αυτό το νοσοκομείο έδωσε σε μία από τις αίθουσες των χειρουργείων το όνομα των τριών κοριτσιών του Ιζελντίν. Πρόκειται για ένα χώρο που είναι στο επίκεντρο του παλαιστινιακο-εβραϊκού προβλήματος και σύγκρουσης. Η Γάζα, παρά την το πρόβλημά της δεν λαμβάνει την αναπτυξιακή βοήθεια και τη βοήθεια ανασύστασης και ανοικοδόμης που θα έπρεπε. Ε, πέρα από το πεπρωμένο αυτής της περιοχής, ε, θα ήθελα να μιλήσω για την πορεία αυτού του ανθρώπου. Τον περασμένο Μάρτιο, ε, ο, ο κ. Πέτερν και εγώ τον συναντήσαμε όταν ήρθε στο Κοινοβούλιο. Και θα το πω με κάθε σοβαρότητα αυτό που λέω. Ποτέ ως βουλευτής δεν συνάντησα έναν άνθρωπο ο οποίος με έκανε σχεδόν να κλάψω, χάρη στο μεγαλείο του, χάρη στον τρόπο με τον οποίο αντιδρούσε στην προσωπική του αυτή θλίψη και στο ε, προσωπικό του δράμα. Όταν του, ε, τον ρώτησα με τι δύναμη μιλάτε για την ε, φιλία, για την συμφιλίωση μετά την τραγωδία αυτή την προσωπική, μου έλεγε σε μένα που είμαι αγνωστική στρία ότι το κάνω γιατί έχω πίστη. Ε, πίστη στο, σε ένα Ισλάμ μετριοπαθές. Ε, ένα Ισλάμ που δυσκολεύεται να βρει την πορεία του στη Γάζα. Γιατί η Γάζα πέρα από τη Χαμάς γνωρίζει και άλλες εξτρεμιστικές ομάδες πιο φονταμενταλιστικές από τη Χαμάς και πιο εγκληματικές συχνά. Επομένως, εάν κρατήσουμε αυτή την υποψηφιότητα του Ιζελντίν, όχι μόνο προωθούμε την ανεξιθρησκεία, την ειρήνη, την αγάπη και τη συμφιλίωση των λαών, αλλά νομίζω ότι δικαιώνουμε έναν άνθρωπο που χρησιμοποίησε την προσωπική του τραγωδία ως σημαία ειρήνης. Πηγαίνει παντού, θα, θα δημιουργήσει και ένα ίδρυμα στη Γάζα για τα νέα κορίτσια ε, και για τη γυναίκα του που πέθανε πριν τρεις μήνες και στη μνήμη των κοριτσιών του, ούτω ώστε τα νέα αυτά κορίτσια να έχουν ένα μέλλον, ένα μέλλον διαφορετικό από τα δικά του. Μιλάω με πραγματική συγκίνηση και ελπίζω να δώσετε μεγάλη προσοχή σε αυτήν την υποψηφιότητα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Απομένει ένα λεπτό για την κυρία Κιλ Νίλσεν. Η ομάδα των Πρασίν θα υποστηρίξει το Memorial, αλλά μερικοί από εμάς θα ήθελαν να υποστηρίξουν τον ε, δόκτωρα Αμποελάης. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε να κάνουμε έναν υψηλό συμβολισμό για αυτό το γυναικολόγο εξαιτία της κατάστασης των παιδιών που υποφέρουν ιδιαίτερα στην Παλαιστίνη μιλήσαμε και είπαμε ότι 300 παιδιά πέθαναν κατά τις 22 ε, μέρες πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Μεταξύ των αμάχων είχαμε ε, να κάνουμε με πάνω από 300 παιδιά που σκοτώθηκαν. Επίσης τα παιδιά υποφέρουν ιδιαίτερα διότι φυλακίζονται. 300-400 παιδιά βρίσκονται συστηματικά στις Ισραηλινές φυλακές. Θα ήθελα να επιμείνω σε, αυτό το, σε αυτή τη σημαντική πτυχή, δηλαδή το πόσο υποφέρουν αυτά τα παιδιά και αυτός ο γυναικολόγος φέρνει στον κόσμο παιδιά από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Νομίζω ότι αποστέλουμε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προς τους νέους άνδρες και γυναίκες που φέρνουν παιδιά στον κόσμο και πιστεύουν ότι πάντα υπάρχει ελπίδα να αποκατασταθεί η ειρήνη σε αυτή την περιοχή και που αναθέτουν σε περχόμενες γενναίες αυτό το καθήκον. Αυτό θα ήθελα να τονίσω θέλοντας να υπογραμμίσω ότι ο δόκτωρ Αμπουελάης δεν ε, περίμενε να πεθάνουν οι κόρες του για να ε, φτάσει σε αυτόν τον αγώνα, διότι τον ε, διεξάγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε την κυρία Κιλ Νίλσεν. Μπορούμε τώρα να περάσουμε την επόμενη υποψηφιότητα, το Ίδρυμα Βισέντε Φερέρ. Η πρόταση έχει γίνει από 39 βουλευτές και τον κύριο Περέγιο, ο οποίος έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποστηρίζω την πρόταση αυτή που έχουν ε, δεχτεί 40 άλλοι βουλευτές από τους σοσιαλιστές και δεν μιλάμε για μία μη κυβερνητική που προάγει αναπτυξιακό έργο. Προβάλλουμε μία πρόταση μίας οργάνωσης ε, προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μειονοτήτων. Των μειονοτήτων που βρίσκονται στο περιθώριο σε ε, και εδώ μιλάω για τους, για τους ανέγγιχτους, για την κάστα των ανέγγιχτων και ιδιαίτερα τις γυναίκες, διότι ανήκουν σε αυτή την πιο περιθωριακή κάστα. Πρόκειται για μια οργάνωση η οποία μιλά για τα οικονομικά και κοινωνικά καθώς και πολιτισμικά δικαιώματα που είναι εντάσσονται στα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να έχουν στέγη, υγεία και τρόφιμα. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια ανθρώπων που δεν πληρούν αυτούς τους όρους έτσι ώστε να βοηθήσει όλους τους περιθωριοποιημένους αυτό το Ίδρυμα, διότι απλούστατα γεννήθηκαν σε αυτόν τον κόσμο. Μιλάμε για μια μεγάλη δημοκρατία. Είναι γεγονός στην Ινδία. Πολλές φορές μιλάμε για έλλειψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλές φορές ξεχνάμε να κοιτάξουμε τις ε, δημοκρατίες. Υπάρχει ελευθεροτυπία, ελευθεροστομία, αλλά πολλοί δεν έχουν ούτε στέγη, ούτε υγεία και ούτε τροφή. Το δικαίωμα στην τροφή, στην διατροφή είναι το, η πιο βασική ελευθερία για να μπορέσουμε μετά να δώσουμε μάχη για την, ε, ε, για τις άλλες ελευθερίες. Μιλάμε για μια μεγάλη δημοκρατία, την Ινδία. Οι οικονομικές, ε, κοινωνικές και πολιτισμικές ελευθερίες φαίνεται ότι δεν θεωρούνται τόσο ανθρώπινα δικαιώματα, δεν εντάσσονται εκεί. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι η πρόταση αυτή πληρεί όλους τους όρους υποψηφιότητας για αυτό το βραβείο και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μιλάμε για, μια, ε, για ένα εγγενές καθήκον, δηλαδή την υπεράσπιση ε, μιας κοινωνικής τάξης που είναι περιθωριοποιημένη. Γεννήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς να τους συμβουλευτεί κανείς σε έναν μακρινό τόπο όπου οι άνθρωποι δεν έχουν ίσα δικαιώματα με τους υπόλοιπους. Όταν μία οργάνωση στην ουσία μιλά όχι μόνο για αυτά τα δικαιώματα, αλλά και για το αυτοδίκαιο αυτών των δικαιωμάτων, ιδιαίτερα μίας περιθωριοποιημένης κατηγορίας, θα πρέπει να την χάνει της δικής μας υποστήριξης. Θα πρέπει να μιλήσουμε λοιπόν για δικαιώματα τα οποία είναι αναφέρετα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο ιδρυτής πέθανε λίγο καιρό πριν, αλλά δεν ζητάμε να απονεμηθεί αυτό το βραβείο στο όνομά του, αλλά σε ολόκληρο το Ίδρυμα, διότι εκπροσωπεί τις περιθωριπμένες μειοψηφίες στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου. Ευχαριστούμε τον κύριο Περέγιο. Περνάμε στην τρίτη υποψηφιότητα, τον κύριο Νταβίτ Ισάκ Η κυρία Εύα Μπρίτε Σβένσον έχει υποστηρίξει αυτή την υποψηφιότητα, δηλαδή υποστηρίζεται από την ΚΟΕ καθώς και τον κύριο Όλε Σμιτ και 31 άλλους ε, υποστηρίκτες. Κύριος Μάγιαρ θα παρουσιάσει την πρόταση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Νταβίτ Ισακ είναι ερυθρέος δημοσιογράφος, συγγραφέας και δραματουργός και ε, έχει αναλάβει αγώνα για την ανεξαρτησία της χώρας του και για τις ελευθερίες της Ερυθρέας. Μία Ερυθρέα η οποία κλειδονίζεται και αποζητά την ανεξαρτησία της στην πρόσφατη σύραξη με την Αιθιοπία. Ο Νταβίτ Ισαάκ κρατήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 2001 διότι στο, στον τύπο δημοσίευσε ένα άρθρο για τις, ε, για τις ελευθερίες στην Ερυθρέα το 2000 που υπερασπίστηκαν πολύ και σήμερα κρατείται ακόμα χωρίς να έχει απονεμηθεί δικαιοσύνη. Και αυτή η δραματική κατάσταση αποτέλεσε αντικείμενο αντίδρασης τον ε, Ιανουάριο το 2009. Εμείς ζητήσαμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την άμεση απελευθέρωσή του και ο τότε πρόεδρος, ο κύριος Πέτερινγκ, απέστειλε μία επιστολή στον πρόεδρο της Ερυθρέας, όπου εξέφρασε την βαθύτατη ανησυχία του για την κλονισμένη υγεία του Νταβίτ Ισάκ και ζήτησε βεβαίως την άμεση απελευθέρωσή του. Ο Νταβίτ Ισαάκ το 87 ήταν πρόσφυγας εδώ στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στη Σουηδία. Ζήτησε να πολιτογραφηθεί ως Σουηδρό στο 92 και γι' αυτό μιλάμε για ένα πολίτη με διπλή υπηκότητα. Ο Νταβίτ Ισάκ ε, εκπροσωπεί την κλειδονισμένη Αφρική η οποία προσπαθεί να προωθήσει ελευθερίες, αλλά δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με καθεστώτα τα οποία στυλιτεύουν όλους τους υπερμαχόμενους των ελευθεριών. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα ήταν ε, πολύ σημαντικό να απονεμηθεί το βραβείο Ζαχάροφ σε αυτό τον υποψήφιο, διότι είναι ειδικό πολίτης, δηλαδή η κατάστασή του είναι ιδιάζουσα αλλά εκπροσωπεί και τους Αφρικανούς ε, και Αφρικανούς πολίτες διότι πρόκειται για μια περιοχή που δεν έχει βασικές ελευθερίες. Χωρίς να σημαίνει ότι υποτιμώ τις άλλες υποψηφιότητες θεωρώ ότι ο Νταβίτ Ισακ πληρεί όλους τους όρους για την απονομή του βραβείου αυτού. Ευχαριστώ κύριε Μάγερ είπατε, το, αναφερθήκατε στο γεγονός ότι ο πρόεδρος Πέτεριν είχε παρέμβει σε επίπεδο κυβέρνησης Ερυθρέας και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη διότι ο πρόεδρός μας έδρασε θαραλέα. Ο κύριος Πέτεριν είναι παρόν και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ε, Μαριάμ Λαμιζάνα είναι η επόμενη ε, υποψήφια έχει προταθεί από τον Φρανσέσκο Φρανσέσκο Σπερώνη, εξ της ομάδας της Ευρώπης της Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Ο κύριος Προβέρα θα παρουσιάσει την υποψηφιότητα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά θα παρουσιάσω αυτή την υποψηφιότητα. Τη θεωρώ εξαιρετικά σημαντική. Γιατί η Μαριάμ Λαμιζάνα ασχολήθηκε και ασχολείται ακόμα με ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θλιβερό σε ορισμένες αφρικανικές χώρες. Είναι μια γυναίκα η οποία ε, ασχολήθηκε με διάφορα κοινωνικά και πολιτικά θέματα και τομείς και είχε τέτοια αξιώματα, αλλά μάχεται και μαχήθηκε στο παρελθόν κατά των ακροτηριασμών των γεννητικών οργάνων των γυναικών. Μία πρακτική που δεν έχει ε, καμία θρησκευτική δικαιολογία, αλλά που την υφίστανται πάρα πολλά κορίτσια. Περίπου 140.000 γυναίκες ε, αφορά αυτή η πρακτική, με βάση μια έρευνα που έγινε. Και περίπου 3 εκατομμύρια γυναίκες το χρόνο κινδυνεύουν να ακροτηριαστούν ε, αυτός ο κριτισμός μπορεί να έχει και πολύ σοβαρές συνέπειες στην υγεία τους. Αυτή η πρακτική γίνεται χωρίς να δοθεί καμία προσοχή στην ε, αντισηψία. Επομένως, οι συνέπειες συχνά είναι πάρα πολύ σοβαρές και σε ορισμένε περιπτώσεις τα κορίτσια ή οι έφηβοι πεθαίνουν κατά τη διάρκεια αυτής της επέμβασης. Η Μάρια Λαμιζάνα είναι Υπουργό Κοινωνική Πρόνοια και Εθνική Αλληλεγγύη στην κυβέρνηση τη Μπουρκίνα Φάσο. Και είναι πρόεδρος μιας εθνικής, μιας διαφρικανικής επιτροπής που καταπολεμά τους ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων των γυναικών. Αυτή η επιτροπή ε, εκπροσωπούσε 20 χώρες αρχικά. Σήμερα εκπροσωπεί 28 αφρικανικές χώρες και συμμετέχουν 15 ε, δυτικές χώρες μέχρι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Νέα Ζηλανδία. Ε, η κοινωνική δράση, περισσότερο από πολιτική δράση της Μαριά Μουλαμιζάνα, έδωσε και πολλά πρακτικά αποτελέσματα. Γιατί στην Πουρκίνα Φάσο η πρακτική αυτή των ακροτηριασμών των γενετικών οργάνων μειώθηκε πολύ σημαντικά δείχνει πραγματικά μια τάση ύφεση, κάμψης, κάτι που είναι πολύ θετικό. Τελειώνοντας, θα να σας πω ότι υπάρχει και κάτι άλλο που θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Δεν πρόκειται μόνο για μια δράση για τη σωματική ακαιρεότητα των ατόμων, αυτή η δράση της Μαρία Λαμιζάν, αλλά μια δράση για τα δικαιώματα των γυναικών. Θέλει να αφυπνίσει τις γυναίκες για τα δικά τους, γύρω από τα δικά τους δικαιώματα όχι μόνο από ιατρικής άποψης, αλλά και από πολιτιστικής και από κοινωνικής άποψης. Είναι ένας αγώνας εξαιρετικά σημαντικός, αν θέλουμε να υπάρξει ένας πιο δίκαιο κόσμος, ο οποίο εξελίσσεται και δίνει ισότητα και στα δύο φύλλα. Το βραβείο Νόμπελ συνήθως ανταμείβει εκείνους που ασχολούνται με και υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά των πολιτικών καταπιέσεων. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται για μια πολιτική καταπίεση, είναι μια πολιτιστική καταπίεση κατά του γυναικείου φίλου που καταπιέζει και παραβιάζει το δικαίωμα στη φυσική ακεραιότητα. Το να ανταμείψουμε αυτή τη γυναίκα, το να τη βραβεύσουμε, το να δείξουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τη βούληση του Κοινοβουλίου ότι υποστηρίζει μια, ένα τόσο δίκαιο αγώνα, και ευγενή αγώνα, νομίζω ότι μπορεί να συνεισφέρει στο να δημιουργήσει στα ενδιαφερόμενα κράτη, εκείνα που, γνωρίζουν αυτό το φαινόμενο, ένα νέο δίκαιο και μπορεί να προωθήσει νομοθεσίες που καταργούν αυτή την πρακτική. Και επίσης βοηθάει στο να υπάρξει μια θύπνιση για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν καλώ τους συναδέλφους, καλώ τους βουλευτές να υπερψηφίσουν και να υποστηρίξουν αυτή την, την υποψηφιότητα. Ευχαριστώ κύριε Προβέρα. Ευχαριστώ κύριε Προβέρα για την ε, παρουσίαση αυτού, αυτής της υποψηφίου. <clears throat> Έχουμε κατόπιν ε, μία πρόταση για την ε, κυρία Λουτμίλα Αλεξέγεβα, τον κύριο Λέγκορλοφ και τον κύριο Σεργέη Κόβαλεφ που εκπροσωπούν την οργάνωση Memorial καθώς ε, και για... Ε, συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση και όλοι οι άλλοι Ρώσοι ακτιβιστές ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πρόταση είναι της κυρίας Ρεμπέκα Χάρμς και του κυρίου Ντάνιελ Πεντή, εξ ονόματος ομάδας των Πρασίνων της Ευρωπαϊκής Ελεύθερη Συμμαχίας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Χάρμς για να παρουσιάσει τους υποψηφίους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η πρόταση που κάναμε και που είναι κάπως πιο γενική, θα ήθελα να την αιτιολογήσω λόγω μιας συζήτησης που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Η Γερμανία συζητάει εδώ και αρκετό καιρό, όλο και περισσότερο φέτος, ότι ε, έχουν περάσει 20 χρόνια από την επανένωση της Γερμανίας. Ακριβώς ε, πριν 20 χρόνια από σήμερα, ε, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Γερμανίας απευθύνθηκε στους στους ε, πρόσφυγες από την ε, Τσεχία και έτσι απευθύνθηκε σε αυτού του ανθρώπους ε, και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία της Επανένωση. Γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Θα πρέπει όμως να λυπούμαστε όταν βλέπουμε το σύνολο της Υπήρου και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών δικαιωμάτων στην Υπηρώ μα πολιτική μου ομάδα πάντα ήταν υπέρ του όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς εδώ και ε, οι πολίτες στα κράτη-μέλη να έχουμε καλές σχέσεις ε, με την Ρωσική Ομοσπονδία. Δεν βρίσκουμε όμως σωστή πάντα την, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην Ρωσία καθώς και στις χώρες του Καυκάσου. Δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και Πιστεύουμε ότι ακριβώς επειδή η προσπάθεια για σταθερότητα και ασφάλεια στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Υπήρου είναι σημαντικό θέμα και είναι σημαντικό θέμα και για την Σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου, γι' αυτό στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να στηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους ακτιβιστές, ε, στα, ε, ε, τους ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ρωσία και στις χώρες του Καυκάσου. Η, η δολοφονία της Άννα Πολικόφσκα καθώς και της Νατάλια Στεμίροβα, θα έπρεπε να μας αποσχολήσουν ιδιαίτερα και γι' αυτό θα θέλαμε φέτος το βραβείο Ζαχάροφ να απονεμηθεί σε υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και στην οργάνωση Memorial που αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τη σπονδυλική στήλη των εργασιών των ε, ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία. Θα θέλαμε με το βραβείο αυτό να τιμήσουμε την κυρία Αλεξέγεβα που είναι μία από τις πιο γνωστές ακτιβίστριες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία. Πιστεύω ότι πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα τη δουλειά της. Ξεκίνησε ήδη επί σοβιετικού καθεστώτος, τότε που χρησιμοποιόταν το σύστημα των Κούλακ και είχε τότε το θάρρος στην τόλμη να μιλήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ε, ανθρώπων αυτών που εργάζονται σε αυτά τα στρατόπεδα εργασίας μαζί με τον ε, Ζαχάροφ ε, μίλησε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και βλέπει την ανάγκη να συνεχίσει τη δουλειά αυτή ε, και στη σημερινή Ρωσία. Ο κύριος Κοβάλεφ το 1996 ίδρυσε μια επιτροπή το 1969 ίδρυσε μια οργάνωση για την πρόσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, που σκοπό είχε να παρακολουθεί ε, πώς ε, εφαρμόζονται στη Ρωσία τα αποτελέσματα της πράξης του Ελσίνκη. Στα πλαίσια λοιπόν της πράξης αυτής του Ελσίνκη πιστεύω ότι αξίζει να απονεμηθεί στον κύριο Κοβάλεφ το, το βραβείο αυτό. Πιστεύω ότι ως πρόσωπο πρέπει να του Πρέπει να του απονεμηθεί το βραβείο και η οργάνωση Memorial με το ιστορικό της, με τη δουλειά που κάνει αυτή τη στιγμή που στη Ρωσία θα πρέπει να λάβει το χρηματικό βραβείο. Με πρόσκληση των προσώπων αυτών όμως και τονίζοντας τη δουλειά των ανθρώπων αυτών και τους κινδύνους ε, που αντιμετωπίζουν, πιστεύουμε ότι Θα τονίσουμε την ε, σημασία του βραβείου αυτού και θα συμβάλλουμε σε μια πιο ασφαλή ήπειρο. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Χάρμς. Έχουμε μία ακόμα υποψηφιότητα που συνδέεται με την οργάνωση Memorial. Ο κύριος ε, Σάριος Βόλσκι και 59 άλλα μέλη πρότειναν την υποψηφιότητα αυτήν. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν ο κύριος Σάριος Βόλσκι θέλει να παρουσιάσει την υποψηφιότητα της οργάνωσης ε, Memorial. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να τονίσω ότι ο ίδιος ο Ζαχάροφ ήταν επικεφαλής ε, της οργάνωσης Memorial. Δεύτερον, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τα όσα είπε η συνάδελφος Ρεμπέκα Χάρμς. Και μάλιστα οι δύο αυτές προτάσεις θα πρέπει να συγχωνευτούν, οι δύο αυτές υποψηφιότητε. Κυρία Χάρμς, και ε, συζήτησα, μαζί σας και με τον ε, κύριο Κον Μπέντιτ ε, την υποψηφιότητα αυτή, καθώς και με άλλους συναδέρφους, διότι είναι ε, διακομματική η πρόταση αυτή. Προτείνουμε λοιπόν να δώσουμε στον Σεργέη Κοβαλόφ, τη Λιουτμίλα Αλεξέγεβα και τον Ολέγκ Όρλοφ το βραβείο αυτό η πρόταση της ε, κυρίας Χάρμς είναι ε, για τους τρεις αυτούς ανθρώπους και όλους τους άλλους Ρώσους ακτιβιστές. Όλοι οι άλλοι Ρώσοι ακτιβιστές είναι η οργάνωση Memorial. Ε, προτείνω λοιπόν να δοθεί στην οργάνωση το βραβείο αυτό, αλλά να προσκληθούν τα, τα τρία αυτά πρόσωπα και να δώσουμε, για να παραλάβουν το, το βραβείο εξ ονόματος της ομάδας. Είναι πολύ σημαντικό το βραβείο Ζαχάροφ, ε, καθότι Παρότι όλοι οι σημερινοί υποψήφοι ε, αξίζουν ένα τέτοιο βραβείο, θα πρέπει να επιλεγεί ο υποψήφιο ανάλογα με τι ε, προτεραιότητε ε, του Κοινοβουλίου. Φέτο έχουμε την ευκαιρία να επιλέξουμε υποψήφιο που όχι μόνο πλήρει τα κριτήρια, αλλά που χρειάζεται και τη δουλειά μα για να συνεχίσει τις, τη δουλειά του σε κάποιε περιφέρειε κλειδιά άμεση γειτονία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στο άρθρο 2 του κανονισμού μας ε, αναφέρονται οι τομείς στους οποίους θα πρέπει να ε, δρουν υποψήφοι και ο υποψήφιος αυτός επληρεί όλα τα κριτήρια αυτά με τρία είδη εργασία ε, πλήρη τα κριτήρια αυτά η Memorial, ε, ε, διατηρώντας την ιστορική μνήμη, με δημοσιεύσεις, με κοινωνική εργασία προς τα θύματα, προς πρόσφυγες, καθώς και ε, πολεμώντας για ίσα δικαιώματα για τις ε, μειονότητες ε, και τρίτον εξετάζοντας την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πρώην σοβιετικά κράτη. Η μη κυβερνητική αυτή οργάνωση εξετάζει την κατάσταση σε κάποιες ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές όπως είναι το Αζερβαϊτζάν, το Τζικιστάν, Μολδαβία, η Βόρεια Οσετία, η Γκουσετία και Ρωσία και ιδιαίτερα Τσετσενία ο χάρτης ε, της Memorial θα μπορούσε να αποτελεί αντίγραφο των ε, προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον εξωτερικό τομέα. Προώθηση της δημοκρατίας με βάση το κράτος δικαίου. κοινωνική επαγρύπνηση, η πρόθεση της αλήθειας όσον αφορά το ιστορικό παρελθόν και αυτό σημαίνει ότι αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση ουσιαστικά εφαρμόζει τους δικούς μας στόχους, τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους και τους στόχους μας ε, όσον αφορά την ε, πολιτική μας ε, στην Ανατολή. Η Memorial είναι φυσικός σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εταίρος αυτός όμως απειλείται. Στο ψήφισμα του 2008 το Κοινοβούλιο μας καταδίκασε το γεγονός ε, ότι έγινε ε, επιδρομή στα γραφεία της Memorial από τις αρχές ε, και κατασχέθηκαν τα αποτελέσματα 20 ετών εργασίας. Φέτος ε, οι ακτιβιστές ε, της ε, Memorial μας λένε ότι η Νατάλια Στεμίροβα βρέθηκε νεκρή και η έρευνα έχει αναβληθεί για δύο μήνες. Έχει ανασταλεί για δύο μήνες και η Memorial έχει αναστείλει τις εργασίες της στην περιοχή αυτή για να προστατεύσει τη ζωή των συνεργατών της σε δύο εβδομάδες ε, το δικαστήριο ε, κατόπιν αίτησης ε, του εγγονού του Στάλιν θα επανεξετάσει την υπόθεση. Θα πρέπει να ενεργήσουμε. Ας αδράξουμε την ευκαιρία αυτή του βραβείου Ζαχάροφ που αποτελεί πολύ σημαντικό εργαλείο της, του Κοινοβουλίου μας να συμβάλλουμε στον αγώνα αυτόν. Ναι, μπορούμε να συμβάλλουμε και ναι, είναι η ηθική μας υποχρέωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σάριος Βόλσκι, για αυτή την πλήρη παρουσίαση της υποψηφιότητας του Memorial. Έχουμε τώρα την υποψηφιότητα του δόκτωρα Ντενί Μουκουβέγγε, που θα την παρουσιάσει ο Γκί Φερχόφστατ από την ομάδα των φιλελεύθερων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει ο κύριος που θα παρουσιάσει τελικά την ε, υποψηφιότητα. Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω το σεβασμό για όλους αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοσίων ελευθεριών. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είδα τη μέρα όπου αναφέρθηκε το όνομα του Σοργέη Κοβάλοφ και του Μεμόριαλ. Γιατί μιλάμε για έναν μεγάλο ουμανιστή και υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, που πραγματικά ήταν στο ύψος ε, των ε, απαιτήσεων του βραβείου Ζαχάρου. Τώρα έχω το προνόμιο να σας παρουσιάζω την επιλογή της ομάδας μου. Κάποιον ο οποίος κέρδισε την ψήφο μας. Είχαμε 10 υποψήφιους και ψηφίσαμε ηλεκτρονικά στο ίντερνετ. Η τρίτη επιλογή του, της ομάδας των φιλελεύθερων, ο δόκτωρας Ντένις Μουκβέγγε. ο συγγραφέας των μονολόγων της, του γυναικείου κόλπου ε, μίλησε ε, θαυμάσια για το πρόβλημα που υπάρχει στο Κονγκό ε, όπου δεκάδες χιλιάδες γυναίκες πέφτουν θύματα βιασμών. Ο δόκτρος Ντένις Μουκβέγγε είναι αυτός που ειδικεύεται στην επανορθωτική χειρουργική των γυναικείων γεννητικών οργάνων στο Κονγκό και έχει αφιερώσει τη ζωή του στην παροχή βοήθειας στις δεκάδες χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια του Κονγκό που πέφτουν θύματα ομαδικού βιασμού και σοβαρή σεξουαλική κακοποίησης. Από την ε, δημιουργία του νοσοκομείου του Πάντζη το 1989 έχει ε, χειρουργήσει πάνω από 21.000 γυναίκες και παιδιά. Ε, τα όσα κάνει ο κύριος Ντένις Μουκβέγγε είναι όλο και πιο δύσκολα, γι' αυτό προσπαθεί να ε, καταρτήσει νοσοκόμες. Το Δεκέμβριο του 2008 και στις αρχές του 2009 ο δόκτορας ε, έλαβε διάφορα διεθνή βραβεία σε αναγνώριση της δουλειάς του ε, για υπέρ χιλιάδων θυμάτων κακοποίησης. Ε, έλαβε και το βραβείο του ΟΗΕ ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το βραβείο Ούλοφ Πάλμε ε, για την πρόθεση της ειρήνης. Και επίσης ένα ίδρυμα της Νιγηρίας τον ονόμασε Αφρικανό της, του 2008. Ο δόκτρος Μουκβέγκε και άλλοι εργάζονται για να καταπολεμήσουν αυτή την επιδημία της βίας στο Ανατολικό Κονγκό. Εκεί χρησιμοποιείται συστηματικός βιασμός γυναικών και παιδιών σαν τρόπος ε, τρομοκρατίας και εκτοπισμού των αμάχων. Νομίζω ότι η ομάδα Άλντε υπέδειξε έναν ε, διάσημο ουμανιστή, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με μεγάλη χαρά σας το παρουσίασα και καλώ τους συναδέλφους να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά του. Ευχαριστούμε κύριε Ραντόνσκης για αυτή την παρουσίαση. Ε, Πρόκειται για την υποψηφιότητα του κυρίου, υπέρ του κυρίου Μουκβέκε. Η επόμενη υποψηφιότητα είναι υπέρ του ευαισιμότατου του Γκουιεν Βαν Λί. Προτείνεται από τον κύριο Μικαέλα Γκάλερ και 44 άλλους. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκάλερ για να μας παρουσιάσει αυτή την υποψηφιότητα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα θέλω να παρουσιάσω την υποψηφιότητα του ε, Βιετναμέζου ιερέα δεσιμότητα του ε, Γκουιν που είναι 61 ετών αυτή τη στιγμή. Ε, από τη ποινή φυλάκιση 8 ετών ε, στο Ναμχά. Από τη δεκαετία του 70 ε, βρίσκεται σε φυλακή περίπου 17 χρόνια συνολικά για την ε, μη η διαμαρτυρία του κατά της ε, κυβερνητικής πολιτικής και, της, και, του, και για την καταστολή των θρησκευτικών δικαιωμάτων. Τον Σεπτέμβριο του 1977 καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 ετών, διότι δημοσίευσε δύο ε, ε, κείμενα του ε, Αρχιεπισκόπου Βανχέη που αναφέρεται στην ελευθερία άσκησης των θρησκευτικών δικαιωμάτων. Απαγορεύτηκε να ασκεί το επάγγελμά του, δεν τήρησε αυτήν την προϋπόθεση και τον ε, Μάιο του 1983 ε, ε, φυλακίστηκε σε 10 έτη φυλάκισης και τον Ιούλιο του 1992 απελευθερώθηκε πάλι. Κατόπιν βρισκόταν υπό αστυνομική εποπτεία και αγωνίστηκε για, για την ελευθερία έκφρασης και άσκησης των θρησκευτικών δικαιωμάτων. Συμμετείχε σε ακρόαση της 16 Μαΐου στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Την επόμενη μέρα συνελήφθηκε και πάλι και τον Οκτώβριο του 2001 ξανακαταδικάστηκε σε φυλάκιση 15 ετών. Λόγω διεθνούς πίεσης ε, απελευθερώθηκε και το 2006 μαζί με άλλους ε, συγγραφείς δημοσίευσε το Μανιφέστο για την Ελευθερία και Δημοκρατία στο Βιετνάμ. Ε, η ομάδα αυτή ονομάστηκε Ομάδα 8406. Μαζί με άλλους ε, ιερείς το 2006 δημοσίευσαν το πρώτο τεύχος περιοδικού που λέγεται Ελεύθερη Έκφραση και το 2000, τον, 8 Σεπτεμβρίου 2006 συμμετείχε στην ίδρυση του Προοδευτικού Κόμματος ε, του, του Βιετνάμ. Το 2007, λόγω του μανιφέστου, ξανακαταδικάστηκε σε 8 επιπλέον έτη φυλάκισης. Κατά τη διάρκεια της ε, δίκης, βιντεοσκοπήθηκε και δημοσιεύτηκε στο ίντερνετ ε, μια, ένα πολύ γνωστό απόσπασμα όπου προσπαθεί να φωνάξει ένα αντικομμουνιστικό σύνθημα ε, ενώ ο αξιωματικός ε, ασφαλείας του έφραξε το στόμα με το χέρι. Ο Γκούιεν Φανλή στις 2 Σεπτεμβρίου του 2009 δεν συμπεριλήφθηκε στην αμνηστία της κυβέρνησης ε, για κρατούμενους. Ο Υφυπουργό ε, Δημοσίας Ασφάλειας είπε, και το λέω στα αγγλικά, ότι η αμνηστία δίδεται μόνο σε άτομα που προοδεύουν ως προς ε, την παρένταξή τους. Δεν έχει αλλάξει, λοιπόν, επειδή δεν έχει αλλάξει θέση ο κύριος Φανλή, δεν συμπεριλήφθηκε στην ε, αμνηστία. Ε, από το 1993 η Διεθνής Αμνηστία τον έχει υιοθετήσει ως κρατούμενο συνείδησης. Με την υποψηφιότητα θα υποστηρίξουμε όχι μόνο τη δική του μη βίαιη διαμαρτυρία ε, για την δημοκρατία και την ελευθερία έκφρασης, αλλά θα στείλουμε και ένα σαφές μήνυμα προς τις αρχές στο Βιετνάμ και θα στηρίξουμε τις δημοκρατικές δυνάμεις εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκάλερ για την παρουσίαση αυτής της ε, υποψηφιότητας που μιλήσατε υπέρ της υποψηφιότητας του Εδεσιμοτάτου, του Ταντέος Μουγιάν Βανλή. Η επόμενη υποψηφιότητα είναι της ε, Σάντι Νάτρ, εξ ονόματος ε, των Ιρανών που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προτάθηκε από την κυρία Μεριέτσι Σάκε, την κυρία Μπάρμπαρα Λόχ Μπίλερ και 38 άλλα μέλη. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και στην κυρία Σάκε και στην κυρία Λόχ Μπίλερ για να μας ε, παρουσιάσουν την υποψηφιότητα της κυρίας Σάντι Σάκρα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους που υποστήριξαν αυτή την ε, υποψηφιότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την υποψηφιότητα που έγινε και από τους, ε, ε, από τους πρασίνους. Όπως ξέρουμε, το Ιράν, μάλλον ξέρουμε, πώς μεταχειρίζεται τους πολίτες του. Και οι άντρες και οι γυναίκες δεν μπορούν να έχουν ελευθερία έκφρασης. Όλοι διατρέχουν το κίνδυνο βασανιστήριων και να χάσουν τη ζωή τους τη στιγμή που υπερασπίζονται ανθρώπινα δικαιώματα που τα θεωρούμε δεδομένα. Ε, ένα σύμβολο αυτών ε, των ε, βασανιστήριων οδήγησε στο θάνατο της Άγκα που είδαμε όλοι. Το YouTube και το Twitter χρησιμοποιήθηκαν για να δούμε ποια είναι η, η αντοχή του Ιρανικού λαού και η αντίστασή του. Η αντίσταση αυτή οδήγησε σε μαζικές διαμαρτυρίες το καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί μια καθημερινή πραγματικότητα στο Ιράν και αφορά ιδιαίτερα στις γυναίκες. Θα σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Πρόκειται για μια πραγματικότητα όπου εντάσσεται και η Σάντι Σάντρ, γιατί πρέπει να υπερασπιστεί αυτές τις γυναίκες ενώπιον του δικαστηρίου οι γυναίκες όταν ε, λιθοβολούνται ε, στην ουσία ε, την χάνουν διακριτικής μεταχείρισης διότι στην ουσία λιθοβολούνται και στην ουσία θάβονται και θάβονται πολύ βαθύτερα από τους άντρες. Πολλές φορές πριν λιθοδοβολιστούν βιάζονται ομαδικά. Η Σάντι Σάντρ υπερασπίζεται αυτές τις γυναίκες ως, ε, ε δι, ως ε, δικηγόρος. Υπερασπίστηκε αυτές τις γυναίκες ε, οι οποίες κατηγορούνται για δίθεν, ε, για δίθεν εγκλήματα και έχει ταχθεί κατά της θανατικής ποινή και κατά του λιθοβολισμού. Επίσης θεωρεί ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν καλύτερη θέση με βάση το οικογενειακό δίκαιο. Επίσης, η κυρία Σάντρ εξτότοπο έτσι ώστε να εκπαιδεύσει τις γυναίκες σε σχέση με, το, με τα δικαιώματά τους. Και η κυρία ε, Σάντρ έχει φυλακιστεί πολλές φορές. Πιστεύω ότι αν της απονομηθεί το βραβείο Ζαχάροφ θα δώσουμε δύναμη στους ίδιους τους Ιρανούς πολίτες έτσι, να έτσι ώστε να καταδείξουμε και στην ε, Ιρανική κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να φέρεται τόσο απάνθρωπα στις γυναίκες. Ευχαριστώ. Κυρία Λοχμπίλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, στηρίζω την υποψηφιότητα της ε, Σάντι Σάντρ ε, για το βραβείο Ζαχάροφ. Έτσι ε, θα δοθεί για πρώτη φορά το βραβείο σε ε, πρόσωπο από το Ιράν, όπως μόλις ακούσαμε η τόλμη της, η επιμονή της ε, και οι έξυπνες ε, και ε, στρατηγικά και στρατηγικές κινήσεις της κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλα αυτά την κάνουν εξαιρετική υποψήφια για το βραβείο αυτό. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η κυρία Σάτι Σάδρ βρίσκεται υπό, γενική, υπό μόνιμη απειλή. Τον Ιούλιο την ξυλοκοπήθηκε. Εάν απονείμουμε τώρα το βραβείο σε ε, μια Ιρανή, ε, αυτό θα γίνει σε μια χρονική στιγμή που πολλοί ε, Ιρανοί αγωνίζονται για τα δικαιώματα τα οποία υπάρχουν στο Σύνταγμά τους. Διαβάζουμε πολλά σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ε, λίγα διαβάζουμε όμως ε, σχετικά με το πόσο ευρύς είναι οι διαμαρτυρίες κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ε, έχουν κοπάσει οι διαμαρτυρίες αυτές. Είναι μια χώρα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ιστορικό σταυροδρόμι. Για πρώτη φορά τα τελευταία 30 χρόνια μιλάμε για μαζικό κίνημα το οποίο έχει ευρία υποστήριξη σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, σε όλες τις ε, κοινωνικές ομάδες και ιδιαίτερα από τους νέους. Χιλιάδες ε, γυναίκες και άνδρες όλων ε, των ηλικιών βγαίνουν στους δρόμους και διακυβεύουν πολλά, διακινδυνεύουν την ελευθερία τους και την ζωή τους. Εάν απονείμουμε το βραβείο στην Σάντις Άντρα, αυτό θα είναι μήνυμα ένα ορατό μήνυμα ε, σεβασμού, ενθάρρυνσης και αλληλεγγύης προς όλους αυτούς που ε, στο Ιράν αγωνίζονται για το δικαίωμα ε, ελευθερίας της έκφρασης, δίκαιων εκλογών κλπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Την κυρία Λοχμπίλερ. Ακούσαμε την υποψηφιότητα για την ε, κυρία Σάντι Σάντρ. Και τώρα έχουμε τον δέκατο υποψήφιο. Η τελευταία υποψηφιότητα είναι αυτή, η δέκατη. Ε, η Σόνια Αλφάνο και 39 άλλοι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν αυτή την υποψηφιότητα. Κύριε Αλφάνο. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους Θα παρουσιάσω τον Ρομπέρτο Σαβιάνο. Ε, είναι μεγάλη τιμή για μένα, λόγω της ιστορίας του, λόγω αυτού που αντιπροσωπεύει. Αλλά θέλω να σας πω ότι και οι υπόλοιποι υποψηφοί είναι ε, μεγάλου βεληνικούς. Ο Ρομπέρτο Σαβιάνο είναι Ιταλός ε, δημοσιογράφος και συγγραφέας 30 ετών. Έγραψε ένα θαυμάσιο βιβλίο, «Τα Γόμορα». Και αμέσως μετά το βιβλίο αυτό, «Η Καμόρα», και όλη η μαφία τον, η καταδίκασε σε θάνατο. Αυτή τη στιγμή ζει σε ένα υπόγειο και αισθάνεται ήδη νεκρός. Δεν είναι ελεύθερος να μοιραστεί τίποτα ε, με κανέναν άλλο άνθρωπο ε, παρά μόνο κάποια λίγα πράγματα με τους συνοδούς του, με τους αστυνομικούς φρουρούς. Θα ήθελα να σας αναφέρω δύο φράσεις ε, του Ρομπέρτο Σαβιάνου που τις έγραψε μία 13χρονη Σικελή. Γιατί πιστεύουμε ότι όλα αυτά που κάνουμε σήμερα ε, αφορούν τους νέους. Νομίζω, είπε, στις, ε, στα 14 χρόνια μια κοπέλα πέθανε από πυρά. Πέθανε από ένα τραύμα στη σποδηλική της στήλη δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αντιδρούμε σε τέτοιου θανάτου με, με χαμηλωμένα βλέμματα. Αυτό που μας έρχεται στο μυαλό είναι να μιλήσουμε και να ουρλιάξουμε. Αγαπητοί φίλοι, ε, λέγομαι Μόνικα και είμαι 13 χρονών. Ε, ζω στην ε, Σικελία, ε, η οποία συνδέεται με τη ζωή της μαφίας. Εγώ δεν την είδα ποτέ τη μαφία, όμως ακούω να μιλάνε, βλέπω ταινίες και Ακούω άτομα τα οποία μιλάνε για τη μαφία και για τα άτομα που σκότωσε η μαφία. Συχνά στις κηδείες όλη η Ιταλία συγκινείται για τους ε, νεκρούς, αλλά εν συνεχεία τους ξεχνάμε. Στη Σικελία, στην πραγματικότητα, συνηθίζουμε σε τέτοια πράγματα, αλλά εγώ δεν μπορώ να συνηθίσω στην ε, κακία και στο φόβο. Ε, πριν από τρία χρόνια, οι γονεί μου αγόρασαν αυτό το βιβλίο του Σαβιάνου, Τα Γόμορα, αλλά δεν το διάβασα. Είδα όμω την ταινία που εμπνεύστηκε από αυτό το βιβλίο και πραγματικά έμεινα κατάπληκτη από το γεγονό ότι ο Ρομπέρτο έχει καταδικαστεί από την Καμόρα επειδή έγραψε αυτό το βιβλίο. Δεν μπορεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Στα 30 του. Ε, οι μοναδικοί άνθρωποι που μοιράζονται τα, τους φόβους ε, και τις σκέψεις του είναι οι φρουροί του. Είναι δυνατόν να κρύβεται αυτός και όχι οι μαφιόζοι που θέλουν να το σκοτώσουν. Νομίζω ότι αν βραβεύσετε το Σαββιάδο θα δώσετε ένα σημάδι ελπίδα σε εμά τους νέους. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο εμείς οι νέοι θα έχουμε κερδίσει μια μάχη κατά της μαφίας. Ε, και για μια φορά το υπόγειο, η υπόγα αυτή στην οποία ζει ο Ρομπέρτο θα ανοίξει ε, σε μια ακτίδα ελπίδας. Ε, ελπίζω κάποια στιγμή να ζήσει μια φυσιολογική ζωή ο Ρομπέρτο, να παντρευτεί και να μπορέσει να οδηγήσει τα παιδιά του στο σχολείο. Εγώ ε, δεν γνώρισα τον, ε, το δικό μου παππού, ο οποίος σκοτώθηκε από την μαφία. Ελπίζω ο Ρομπέρτο να μπορέσει να συνεχίσει να ζει. Ε, αν βραβεύσει τον ε, Ρομπέρτο Σαβιάνο, θα μας δώσετε μία πνοή ελπίδας. Πολύ ωραία, λέει η κυρία Χαουτάλα. Ακούσαμε τις υποψηφιότητες 10 εξαιρετικών ε, ανθρώπων, υποψήφιοι για το βραφείο Ζαχάροφ, αιτιολογήθηκαν οι υποψηφιότητες. Έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε σύντομα απόψεις. Θα ήθελα να είσαστε λακωνικοί. Έχω τον κύριο Λανσμπέργκης και την κυρία Ντεκάιζερ. Μέχρι να είσαστε, σας παρακαλώ, πολύ λακωνικοί όμως. Thank you, madam. Colleagues, so let me remind to you once more, following Mr. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μετά από τον κύριο Σάρι θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, Νατάλια Εστεμίροβα ε, που ήταν ε, θύμα στην Τσετσενία, σκοτώθηκε λόγω... Πέθανε επειδή οι αρχές καταδίκασαν τις ενέργειες της, όπως είχαν καταδικάσει και τις ενέργειες ε, της Άννα για Η κυρία Εστεμίροβα ήταν η υποψήφια για το βραβείο Ζαχάροφ ε, πριν κάποια χρόνια. Όπως και ο κύριος Ζέρκε Κόβαλεφ. Μετά από συζήτηση μεταξύ των ε, πολιτικών ομάδων δόθηκε το βραβείο σε, ε, στην ομάδα ελεύθερων δημοσιογράφων, ενώ σε αυτούς ε, απενημήθη το ε, μετάλλιο Ρόμπερτ Σούμαν. Η κυρία Εστεμίροβα δεν βρίσκεται πια μαζί μας, ο Σέργεϊ Κόβαλοφ όμως και οι άλλοι δύο είναι, ζουν ακόμα. Η οργάνωση Memorial δεν έχει απαγορευτεί ακόμα, παρότι διώκεται. Ε, έχουν εκδιωχθεί από την Τσετσενία που δείχνει τρομερή διαφορία απέναντι σε τέτοιες ε, δολοφονίες. Έχουμε λοιπόν την μοναδική ευκαιρία να εκφράσουμε την υποστήριξή μας ε, προς τους θαραλέους αυτούς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τέτοιους τομείς. Η, η κοινή υποψηφιότητα της οργάνωσης ε, και κάποιων εξεχόντων προσώπων της οργάνωσης αυτής. Πιστεύω ότι αξίζει την υποστήριξή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λάνσπερκης. Ελπίζω ο κάθε μιλητή να περιοριστεί σε ένα λεπτό αν είναι δυνατόν, διότι έχουμε άλλο ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη μετά από τη συζήτηση αυτή. Η κυρία Κάιζερ. Ένα ενημερωτικό σημείο και ζητώ συγγνώμη που παίρνω τον λόγο. Η ομάδα μου, η σοσιαλιστική ομάδα, δεν, παρουσιάστηκε, δεν παρουσίασε δική της υποψηφιότητα γιατί είχαμε άλλους υποψηφίους. Αλλά καθώς βιαστήκαμε να υπογράφουμε, δεν είχαμε το χρόνο να προσυπογράψουμε την υποψηφιότητα της κυρίας Άντι Σάντρα. Θα ήθελα να το τονίσω για να δείξω και αλληλεγγύη προς τους πράσινους ότι κάποιοι σοσιαλιστές θα υποστηρίξουν τις αντισάντρ. Ευχαριστώ την κυρία Ντεκάιζερ. Ο κύριος Μάουρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπορώ να αισθανθώ ήσυχος, γιατί πραγματικά οι υποψηφιότητες που ακούστηκαν ήταν εντυπωσιακές αν τα πρόσωπα, οι υποψηφιότητες αυτές είναι τόσο μεγάλου βεληνικούς, φανταστείτε πόσο εντυπωσιακό είναι, εντυπωσιακός είναι ο αριθμός των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο. Ακούγοντας ε, λοιπόν τους συναδέλφους, μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι κατάλαβα ότι υπάρχουν σημεία στον πλανήτη όπου σταματάει περισσότερο το βλέμμα μας και η προσοχή μας. Γιατί θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό να γίνονται τέτοιες παραβιάσεις. Παραδείγματος χάρη παρουσίαση που έκανε ο κύριος Γκάλερ. Ε, εδώ και χρόνια ασχολούμαι με το Βιετνάμ. Ε, πάντα θετικά. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται εκεί, βελτιώνεται. Κι όμως νομίζω ότι το βραβείο Ζαχάροφ είναι μια θαυμάσια περίπτωση και ένα θαυμάσιο μοχλός για να θέσουμε την προσοχή όλων σε αυτές τις χώρες, σε αυτά τα μέρη του πλανήτη, όπου υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ, κύριο Σμίτ. Έχει ένα λεπτό. you, I, um, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μία έκκληση υπέρ του δημοσιογράφου Τάβιτ Ισακ. Βρίσκεται στη φυλακή εδώ και 8 χρόνια, από τις 23 Σεπτεμβρίου του 2001. Και Βέβαια είναι πολύ δύσκολη η θέση του, όπως ε, μάλλον γνωρίζουμε, δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι. Είναι ε, πολύ άρρωστος, ε, δεν είχε δίκαιη δίκη και συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, από ό,τι γνωρίζω είναι ο μόνος ο μόνος πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στη φυλακή επειδή ε, του θεμελιώδους δικαιώματος να εκφράζεται ελεύθερα. Πολίτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται 8 χρόνια στη φυλακή στην Ασμάρα και δεν κάνουμε τίποτα. Όχι τίποτα, αλλά όχι αρκετά. Η οικογένειά του στο Γκέτεμποργκ, όπου αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, δεν γνωρίζει τίποτα γι' αυτόν. Το βραβείο Σαγάροφ ε, νομίζω θα τον βοηθήσει, μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωσή του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σμιτ. Να τονίσω ότι και ο κύριος Σαβιάνο είναι υπήκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Μισής Κυρία Μουνίθ, όλες οι υποψηφιότητες που ακούσαμε είναι εξαιρετικές υποψηφιότητες. Ορισμένες μας εγκίνησαν πολύ. Πίσω από αυτές υπάρχουν δραματικές ιστορίες συχνά. Νομίζω ότι είναι όλες αξιοπρεπείς και αξίζουν όλοι το βραβείο. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προωθήσουμε μία υποψηφιότητα που ξεπερνάει το πρόσωπο και που μπορεί να έχει ένα πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, να έχει δηλαδή επίπτωση στις ζωές πολλών ανθρώπων ιδίως για ανθρώπους που βρίσκονται σε δραματικές συνθήκες, που δεν έχουν θεμελιώδη δικαιώματα και που θα πρέπει λοιπόν και θα πρέπει με αυτό το βραβείο να αγγίξουμε περισσότερους από έναν ανθρώπους, παρότι συχνά ε, τα μεμονωμένα άτομα ε, ζητούν, ζουν σε δραματικές συνθήκες. Ακριβώς αυτή η οργάνωση, η Βισέντε Φερέρο, είναι μια οργάνωση που βοηθάει πάρα πολλά άτομα στην Ινδία, μια πολύ φτωχή χώρα. Ακόμα δύο παρεμβάσεις και εν συνεχεία θα πρέπει να κλείσω το, δυστυχώς τον κατάλογο των, των ομιλητών. Ο κύριος Σβόμποντα και ο κύριος Σούλτς. κύριος Σβόμποντα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ δύσκολο να διαλέξει κανείς. Προσωπικά Υποστήριξα την ε, υποψηφιότητα του Παλαιστίνιου γυναικολόγου. Πιστεύω ότι είναι υψή τη σημασίας να δώσουμε ευκαιρία στην ειρήνη. Θα ήθελα όμως να πω ότι η αντιπροσωπεία των ε, σοσιαλδημοκρατών ε, βρέθηκαν στην, στη Ρωσία, στη, στη Μόσχα και συναντήθηκαν με εκπροσώπους της Memorial. Η Memorial κάνει πολύ σημαντική δουλειά και άσχετα από την απονομή του βραβείου, πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τον διάλογο με τη Μεμόρια. Ήθελα να το αναφέρω, ε, διότι θέλω να καταστήσω σαφές ότι η ε, υποψηφιότητα, η απόφαση υπέρ κάποιου δεν αποτελεί απόφαση κατά των άλλων. Ήθελα απλά να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Σβόποτα, πολύ σημαντική παρατήρηση. Και συμφωνούμε απόλυτα. Τελευταία παρέμβαση ο κύριο Σούλτ, παρακαλώ. Μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα με τον προαναλύσαντα κύριο Σφόποτα. Η κάθε μία από αυτές ε, αξίζει το βραβείο Ζαχάροφ, ε, γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να περιοριστούμε ε, στα κριτήρια. Μία ζωή, αγώνα αφενός και αφετέρου να σκεφτούμε και τι πολιτικέ συνέπειε. Η κατασυρωή δολοφονία δημοσιογράφων στην Ρωσία είναι κάτι που διακυβεύει την κοινωνία των πολιτών ε, και πιστεύω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή επιδεικνύουν ε, απίστευτη τόλμη και τώρα και στο παρελθόν ε, υπερασπιζόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ προέρχομαι από την αντίσταση στην Ανατολική Γερμανία. καταφέραμε μια ειρηνική επανάσταση επειδή υπήρξαν αυτοί οι ε, Ρώσοι οι οποίοι ξεκίνησαν ε, την ε, διαδικασία του Ελσίνκη. Πιστεύω λοιπόν ότι ε, αξίζει να, δοθεί, να απονεμηθεί σε αυτούς το βραβείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σούλτς. Πολύ ωραία. Εν είδη σύνοψης και κατάληξης, να σας υπενθυμίσω τη διαδικασία. Θα γίνει μια ενδεικτική ψηφοφορία με βάση ένα short list στις 6 Οκτωβρίου την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Θα γίνει μία συνεδρίαση ε, και κλεισμένων των θυρών και εκεί θα λάβει η χώρα η ψηφοφορία. Εν συνεχεία, η επόμενη φάση, η διάσκεψη των Προέδρων θα ψηφίσει στο Στρασβούργο στις 22 Οκτωβρίου Ο νικητής θα προσκληθεί εδώ στις 14 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο σε μια συνεδρίαση ΑΦΕ, ΔΕΒΕ και Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια μεικτή επιτροπή, στις 14 Δεκεμβρίου. Είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία. γιατί θα συμπληρωθούν 20 χρόνια από την ημερομηνία που ο Ανδρέη Ζαχάροφ θα μας έχει εγκαταλείψει. Η επίσημη τελετή θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο. Η γραμματεία του Κοινοβουλίου θα κάνει ό,τι μπορεί, ούτω ώστε η προσοχή των ΜΜΕ να στραφεί σε αυτό τον νικητή για τη δουλειά που θα έχει επιτελέσει υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι το βραβείο Ζαχάροφ από χρόνο σε χρόνο γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας ευχαριστήσω. Με μεγάλη χαρά άκουσα αυτές τις 10 υποψηφιότητες για το βραβείο Σαχάροφ 2009. Κλείνω αυτό το σημείο προς το παρόν, αλλά έχουμε το σημείο 3 της ημερησίας διάταξης οι επιτροπές μας από κοινού αποφάσισαν να παρουσιάσουν μια προφορική ερώτηση στο Συμβούλιο που αφορά την ε, υποστήριξη της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άφε, τέβε, υποεπιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προφορική ερώτηση και των τριών. Για ποιο λόγο η Σουηδία, που έχει και την Προεδρία στο Συμβούλιο, επιθυμεί να συζητήσουμε την οικοδόμηση της δημοκρατίας, στις εξωτερικές σχέσεις, γιατί θεωρείται μια προτεραιότητα στις εξωτερικές σχέσεις από τη Σουηδία. Η Προεδρία της Σουηδίας θεωρεί ότι πρέπει να έχουμε μια συνεκτική πολιτική, Ένα τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δράσει για να οικοδομήσει ή να προωθήσει τη δημοκρατία ανά τον κόσμο. Και στο Συμβούλιο 16 και 17 Οκτωβρίου Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα συνταχθούν συμπεράσματα για αυτό το στόχο. Ο στόχος είναι με οριζόντιο τρόπο και, στα τρία, και στους τρεις πυλώνες να συζητούμε το πώς μπορούμε να προωθούμε καλύτερα τη δημοκρατία. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε αυτό το κοινό ερώτημα προφορικό ερώτημα. Οι συντονιστές της Επιτροπής ΔΕΒΕ θα υιοθετήσουν ένα κείμενο από ό,τι μου λένε τη Δευτέρα στις 28 Σεπτεμβρίου. Υιοθέτησαν μάλλον ένα κείμενο. Δεν θα ήθελα να μιλήσουμε για τις λεπτομέρειες αυτού του κειμένου. Θα μπορούσαμε από κοινού να συμφωνήσουμε αυτό το προφορικό ερώτημα να το κάνουμε δικό μας, ούτω ώστε να μπει στην ημερήσια διάταξη στην ε, συνεδρίαση του Συμβουλίου. Επομένως, συμφωνείτε να υιοθετήσουμε αυτό το προφορικό ερώτημα. Καμία αντίρρηση, πολύ ωραία. Θα παρουσιάσουμε αυτό το προφορικό ερώτημα στο Συμβούλιο. Σημείο 4, διάφορα. Δεν υπάρχουν σημεία από τα διάφορα. Σας ευχαριστώ. Λύεται η συνεδρίαση.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 1, 2, 1, 2.